Συνάδελφοι, ε, στην ε, ημερήσια διάταξη εμφανίσεται το επόμενο θέμα που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά, στην κυρία ε, Αντρικένε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωπε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που σας βλέπω σήμερα μαζί μας στην αίθουσα της Ελλομέλειας. Είναι ιδιαίτερη σημασία σε αυτή η συζήτηση, διότι είναι ακριβώς η πρώτη συζήτηση πολιτικού χαρακτήρα που κάνουμε από την άνοιξη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας για την Εξωτερική Δράση. Εδώ το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε αύριο βασίζεται στην έκθεση του Συμβουλίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2009, καθώς και τις πολιτικές της Ένωσης σχετικά. Κυρία Άστον, δεν μπορούμε βέβαια να σας θεωρήσουμε υπεύθυνοι για όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο, για όλα τα, όλες τις δράσεις που αναφέρονται στον λόγο έγγραφο, γιατί για την περίοδο 2008-2009 δεν είχατε ακόμη αναλάβει καθήκοντα, όπως και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι έχετε αναλάβει σοβαρότατες ευθύνες. Και πραγματικά από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε τις φιλοδοξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική να τις επιδιώξουμε από κοινού. Κυρία Άστον, εδώ και ένα χρόνο τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Η υπηρεσία τη οποία ηγείστε ε, ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδε τι εργασίε του. Σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο αποστέλει ένα σαφέ μήνυμα προ όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε ότι η νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην υπεράσπιση της δημοκρατίας ε, στον κόσμο και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παντού ανά την Ιφίλιο. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο μέλλον, το μελλοντικό σχεδιασμό του οργανισμού αυτού. Μιλάμε για την τήρηση τη ειρήνη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για διαφορετικέ δομέ όμω με την ε, ίδια αποστολή. Δεν θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να χαθούν ε, από τι προτεραιότητε, από τον κατάλογο προτεραιοτήτων τη υπηρεσία, ούτε από τη δομή του οργανισμού. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν προτείνει στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής να προβλεφθούν λειτουργίες ειδικών απεσταλμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απεσταλμένοι οι οποίοι να εργάζονται εκεί όπου δεν έχει μόνιμες αντιπροσωπείες ή διπλωματικές ε, αντιπροσωπείες η διπλωματικες αντιπροσωπιες η Ένωση. Θα πρέπει να έχουν σαφεί, ξεκάθαρε εντολέ οι άνθρωποι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι χώρε όπου θα αναλαμβάνουν καθήκοντα. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να υπάρχει μια ομάδα επιφορτισμένη με τα θέματα αυτά, καθώ ε, η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι υπέρ μια τέτοια πρωτοβουλία. Στην έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, συζητάται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μία σειρά αποζητήματα. ζητήματα. που αφορούν την κατάργηση της θανατικής ποινής, την εργασία των παιδιών, την καταπολέμηση των βασανιστήριων, την βελτίωση της συνθήκης, των συνθήκων διαβίωσης των γυναικών σε διάφορες χώρες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης και ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Εδώ στην έκθεση αυτή κάνουμε λόγο για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή ο ΙΕ. Ε, μιλάμε και για τη συνεργασία μας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η έκθεση λοιπόν που ετοίμασα ε, στηρίχθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους, βουλευτές, ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι περισσότεροι υπερψήφισαν την έκθεση, κανείς δεν την καταψήφισε και απλώς δύο απήχαν. Σήμερα λοιπόν ήθελα να τονίσω ότι κανένα σημείο δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εγώ ήθελα εδώ να παρουσιάσω δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να με το βραβείο Σαγάροφ στον κύριο Φαρίνια, τον κύριο Γιγέρμο Φαρίνια. Δεν μπορεί όμω να γίνει αυτό, γιατί οι κουβανικέ αρχέ δεν έδωσαν το δικαίωμα στον κύριο Φαρίνια να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων σα θα το λάβετε αυτό υπόψη και θα βρείτε τρόπο ώστε να εκφράσετε κι εσεί τη δική σα την στάση, την θέση και την δυσαρέσκειά μα ε, έναντι των κουβανικών αρχών για αυτή του την ε, δράση. Και για μια άλλη περίπτωση, περίπτωση την οποία αναφέρουμε και στην έκθεσή μα. Σήμερα το ρωσικό ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για μια συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά για άγνωστου λόγου ανεβλήθη η εκδίκαση τη υπόθεση για αργότερα. Μιλάμε για την υπόθεση Μικαήλ Κοντοκοφσκή και του συνεταίρου του, του κυρίου Λεμπεντεφ. Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι δεν υπερισχύει το κράτο δικαίου στη Ρωσία. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε μου, να, κάνετε όλ, να καταβάλλετε όλε τι απαραίτητε προσπάθειε ώστε η δικαιοσύνη να γίνει ένα κανόνα που όλοι ακολουθούν, όχι μια εξαίρεση. Και για τη Ρωσία. Ε, η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα. Ο πρόεδρο Μεντβεντέφ έχει τη διάθεση να εξυγχρονίσει τη χώρα. Αυτή πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και εμεί από την πλευρά μα να τον στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τον ε, λόγο έχει η αντιπρόεδρο κυρία Άστον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Την Παρασκευή είχαμε την ημέρα τη Διεθνή Μέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εκεί λοιπόν προβάλαμε ε, την εργασία ατόμων αλλά και οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο για, κυρίως για όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν ε, την καταπολέμηση, που προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτά τα φαινόμενα. Είχαμε λοιπόν την ε, το Σαβάη Μπράγκ που επιβραβεύτηκε και άλλους που υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Όπως είπα και προηγουμένω. Ε, θεωρώ ότι οι συνάδελφοί μου στις Βρυξέλλες και οι επικεφαλείς ε, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πράξουν το ίδιο. Πριν από έξι μήνες ήμουν εδώ για να σας παρουσιάσω ένα όραμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα θέλω να σας πω πώς ακριβώς προχωρεί η υπόθεση αυτή έκτοτε και τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον με την υποστήριξη της ε, υπηρεσίας του εξωτερικής δράση. Πρώτα απ' όλα όμως είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στη δόκτωρα Αντρικένεν για την έκθεσή της ε, που ταυτίζεται με την έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρουσιάζει το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς μπορούμε να καταστήσουμε την προστασία τους πιο αποτελεσματική. Αυτή είναι μια φιλοδοξία που συμμερίζομαι και εγώ. Οι ε, πράξεις, ε, οι πράξεις που αναλαμβάνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα εμφανίζονται πολύ καλά στην έκθεση. Η χρήση νέας τεχνολογία για την διατήρηση τις ελευθερίες της έκφρασης. Αυτά αναφέρω ενδεικτικά. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την προσπάθεια της κυρίας Αντρικέν για το ότι κατέθεσε πάνω από 400 τροπολογίες σε αυτή την τόσο χρήσιμη και ενημερωτική έκθεση, η οποία καλύπτει ένα τεράστιο πεδίο. Και θα ήθελα να φερθώ σε τρεις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δούλεψε σκληρά για να προωθήσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την, μια κοινή άποψη για τα ψηφίσματα σχετικά με την Γκάζα Φλωτήλα και την έκθεση Κόλστον. Όσον αφορά την τρίτη, ε, τη συνάντηση της Επιτροπής ε, για που ασχολήθηκε με τη Βυρμανία ε, και με την ε, θανατική ποινή. Αυτά όλα πέρασαν με ενισχυμένη πλειοψηφία όπως και το ψήφισμα για το Ιράν και το ψήφισμα για την εξάλληψη της μυσαλλοδοξίας της θρησκευτική. Όπως είπαμε και τον Ιούνιο, ε, ε, άρχισε η αναθεώρηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί συνέβαλαν τα κράτη-μέλη, οι βουλευτές, η κυρία Χάουταλα και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως επίσης και οι κοινωνίες των πολιτών, ΜΚΟ και Ακαδημαϊκή. Ε, τους επόμενους μήνες ζήτησα από τους συνεργάτες μου να λάβουν υπόψη τους τα θέματα που θα προκύψουν και τον καλύτερο τρόπο πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά. Ε, θα υπολογίζω στην προσπάθεια, στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτή την προσπάθεια. Τρίτον, ε, άρχισε ε, κάποιο συντονισμό των πολιτικών που προέκυψαν τα τελευταία δέκα χρόνια και αυτά θα αποτελούν τι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε δύο εργαλεία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχουν και λόγοι γιατί έχει προχωρήσει τόσο καλά η συνεργασία. Όμω είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε απολογισμό και να προχωρήσουμε. Από αυτή λοιπόν την αναθεώρηση βλέπω ότι θα ε, προκύψουν τρει γραμμέ δράση. Πρώτον, η ανάγκη για την Ευρώπη να εκφράζει την άποψή τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τι ε, πράξει μα σε επίπεδο ε, Ηνωμένων Εθνών θέλουμε να βρούμε καινοτόμους τρόπους για να συνεργαστούμε με εκπροσώπους ε, τρίτων χωρών, όπως ε, το κάναμε πάρα πολύ καλά στο ψήφισμα για τη θανατική ποινή. Επίσης, επιθυμούμε ε, και τα δικά μας τα πεπραγμένα να ελέγχονται. Θέλουμε την δική μας την προσέγγιση να την προσαρμόσουμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Άρα δηλαδή τοπικές ε, στρατηγικές αναθεώρηση των πρακτικών μας και βέλτιστη χρήση των εργαλείων που διαθέτουμε. Παραδείγματο χάρη ανταλλαγή πληροφοριών για την προστασία ε, των παιδιών από το ίντερνετ ή της παιδικής εργασίας. Τέλος, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Πρέπει δηλαδή να ενταχθούν σε όλες τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η υπηρεσία εξωτερικής εξωτερικής δράσης όπως επίσης και σε πολλές άλλες πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα. Αυτά λοιπόν ε, θα λάβουν χώρα για να μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούμε αποτελεσματικά ε, να ε, διεκδικούμε τους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η πεμπτουσία της ταυτότητάς μας και είναι στο στον πυρήνα εκείνων που επιδιώκουμε. Θέλουμε λοιπόν τις αξίες αυτές ε, να τις προάγουμε σε ένα πολυμερές επίπεδο και με την υποστήριξη της ε, κοινωνίας των πολιτών. Η χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πάνω από 100 χώρες. Δέκα χρόνια από την πρώτη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τη σύσταση της νέας υπηρεσίας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική μας είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και στοχευμένη το οδηγό αυτό νήμα που διατρέχει όλες ε, τις ε, δράσεις μας ε, είναι εκείνο που καθορίζει και την εξωτερική μας πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε να τελειώσω τον νικητή του βραβείου Ζαχάροφ για τη σκέψη του και την ελευθερία του πνεύματος. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητέ των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ. Ο κύριο Βαϊντερε για ένα μισή λεπτό έχει το λόγο. Η κυρία Βαϊντέρη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Αντρική Ένα για την έκθεση που υιοθετήθηκε σχεδόν ομόφωνα. Επίσης ευχαριστώ την κυρία Άστον για ε, της ε, πλήρη της ε, τοποθετήσεις της. Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο δείχνει σε πόσο κριτική κατάσταση βρίσκονται οι χώρες, ακόμη και χώρες με τις οποίες εδώ και πολλά χρόνια συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία πληρεί μόνο μία από τις έξι ρήτρες που έχουν υπογραφεί Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Νότιο και στην Απχαζία και θα πρέπει να επιληθούν τέτοια σειράξει και γι' αυτό πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας σε τέτοια ζητήματα. Είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να καταβάλει προσπάθειες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν γι' αυτό στην ε, πολιτική για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Καταρχήν θα πρέπει να συστήσουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα που να καθορίζει όχι μόνο τα καθήκοντα αλλά και μια δομή που να μας ε, δίνει μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιθυμούμε. Δεύτερον, αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία μας και σε ορισμένα προσδιορισμένα κριτήρια. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε την άποψή μας επειδή θα σκείται πίεση από τρίτη χώρα ή λόγω οικονομικών συμφερόντων. Τρίτον, πρέπει να έχουμε διαβουλεύσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εγγυηθούμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει αυτό να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και για τη σύναψη σχέσεων μας με τις τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα για την ομάδα των σοσιαλιστών η κυρία Ντεκέισερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ εκτενής και είναι ιδιαίτερα εξαντλητική σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα έχει κάποια μειονεκτήματα ε, όπως ε, παραδείγματος χάρη ότι είναι ιδιαίτερα μακροσκελής ε, ε, αλλά δεν φταίει η συγκήτρια γι' αυτό, αλλά ο τεράστιο αριθμό των ε, τροπολογιών που έπρεπε να συμπεριληφθούν. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Τρικέν. Επίση, φαίνεται εδώ ότι ε, τα ανθρωπίνα δικαιώματα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και συνεπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σα ζητά, κυρία Άστον, ένα ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γενική διεύθυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατάρτιση για το προσωπικό και να υπάρχει και κάποιος ο οποίος να εποπτεύει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις τρίτες χώρες. Αν επιθυμεί το Κοινοβούλιο τέτοιε δομέ δεν είναι για να έχουμε μεγαλύτερη γραφειοκρατία αλλά γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αυτή η ε, έκθεση ε, ουσιαστικά ε, δεν αποτελεί απλώς μια παρήθμιση ε, της φρίκης. Ε, κάνει κάποιες συστάσεις για τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν και για το διάλογο που πρέπει να γίνει. Αντικατοπτρίζεται και ο πλούτος του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτό Εδώ έχουμε ένα σύνολο εργαλείων που μπορούν να συνεισφέρουν για την πρόθεση της δημοκρατίας στον κόσμο. Πρέπει επίσης να πιστούν οι συνομιλητές μας ότι τα ανθρώπινα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν φρένο στην ανάπτυξη και στο διεθνές εμπόριο, ε, δεν αποτελούν ε, ε, κάτι αφηρημένο που θα υπάρχει στις εξωτερικές σχέσεις, αλλά αποτελούν παράγοντα ευημερία και σταθερότητας. Κυρία, ε, εκπρόσωπος πάρα πολύ καλά πήρατε τη σκητάλη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δηλώσατε ε, τη δεσμευσή σας ε, κατά το πρώτο αυτό έτος που ακολούθησε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και εμείς εκ μέρους των φιλελευθέρων για δύο λεπτά ο κύριος Ντόνσκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους ε, για τις τροπολογίες. Εγώ θα συνεχίσω τις προσπαθίες μου για την τελειοποίηση αυτής της έκθεσης. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε αναλάβει ορθά την πρόκληση και Έχουμε λάβει και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό μας επέτρεψε να βελτιώσουμε την έκθεση. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι πρέπει να θετήσουμε την έκθεση αυτή, η οποία αντικατοπτρίζει ορθά τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ζητήσω από τους συναδέλφου ε, να μην σταθούν σε ζητήματα που έχουν ήδη συζητηθεί. Παρ' όλα αυτά, ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές χώρες για τις οποίες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τα προβλήματά τους αλλά πρέπει να μην ε, χάσει την αποτελεσματικότητά της η έκθεση αυτή. Θέλω να αναφερθώ σε ορισμένε τροπολογίες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη εκδοχή. Παίρνουμε τους χάρη ε, κάποια τροπολογία που αναφέρεται στη θανατική ποινή. Ε, μια ουσία πρέπει να πωλείται συγκεκριμένα εισόδικ, πρέπει να πωλείται μόνο για θεραπευτικούς ε, σκοπούς. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να υιοθετήσουμε αυτά που λέμε στην έκθεση του 2007 για το ζήτημα αυτό. Αυτό το έγγραφο δεν αποτελεί απλώς ε, ένα σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών. αλλά κατευθυντήριες γραμμές και για τις χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω οι συστάσεις αυτές να υιοθετηθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για τους πράσινου, η κυρία Χαουτάλα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και εγώ την υπατή εκπρόσωπο στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα και ήθελα να συγχαρώ θερμά την κυρία Αντρικένε για το έργο της. Είναι εξαιρετικό το έργο γιατί δουλέψαμε ως ομάδα και ελπίζουμε ότι σχεδόν ομόφωνα θα εγκριθεί. Και έτσι εγκρίθηκε και στην Επιτροπή για τι Εξωτερικέ Υποθέσει. Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή που φέτο ε, στο φθινόπωρο να συμμετάσχω στι συζητήσει μεταξύ κρατών μελών ε, για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαμορφώσει την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη συνέπεια πιστεύω ότι έχουμε πλέον, ε, είμαστε, έχουμε στα χέρια μας μια αντιμέτωπη, έχουμε στα χέρια μας μια ιστορική στιγμή για να προχωρήσουμε με τις προτεραιότητες της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εσείς αναφέρατε κυρία Άστον. Η δική μου πρόταση θα ήταν η εξής, η διαδικασία αυτή να ε, προκαλέσει τη συμμετοχή των δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων. Γι' αυτό ήθελα να σα ε, συστήσω, αν θέλετε, και στην επικοινωνική σα πολιτική ε, αυτό το χρόνο ε, και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο να οργανώσετε συζητήσει υψηλού επίπεδου σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το θέτει το θέμα αυτό στον πυρήνα τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε τι κατάλληλε υποδομέ σε λειτουργία. Γνωρίζουμε ότι εσεί, είπατε εκπρόσωπο, έχετε αναλάβει δεσμεύσει ε, στο επιτελείο σα ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τη δημοκρατία. και ελπίζουμε να το δούμε αυτό να μεταφράζεται και σε πράξη. Μπορείτε να μα πείτε αν ε, θα εκπληρωθεί η υπόσχεση που δώσετε και στο Κοινοβούλιο το καλοκαίρι. Επίση, σα παρατηρώ θερμά να ε, προχωρήσετε σε απόφαση για να δημιουργήσετε την ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ΚΟΧΟΜ, που να βασίζεται στι Βρυξέλλε. διότι αν θέλουμε περισσότερη συνέπεια, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και αυτή τη μόνιμη δομή. Ε, τέλος, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας προκειμένου να φέρετε σε σύγκληση τα κράτη-μέλη και να κανονίσετε συνάντηση την τελευταία Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή στο Όσλο. Νομίζω ότι χωρίς τις δικές σας έντονες προσπάθειες δεν θα είχε γίνει η συνάντηση αυτή. Ήταν μια πολύ καλή βάση για να συνεχιστεί η εργασία μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε η Ένωση να έχει μια ισχυρότερη, ξε, πιο ξεκάθαρη και πιο αποτελεσματική φωνή παγκοσμίω. Ευχαριστούμε εκ μέρου ε, των συντηρητικών και ευρωπαίων μεταρρυθμιστών Σιμάνσκι για ένα ε, λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι η εισήγηση αυτή είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και θέλω να πω το εξή. Οι χριστιανοί είναι περισσότερο διοκόμενοι ανά τον κόσμο. Τους επιτίθενται, τους δολοφονούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όμως ε, αυτό δεν επισημαίνεται, κανείς δεν μιλάει. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ λίγα κάνει για αυτό το θέμα. Είμαι ευγνώμων σε εσά, Lady Ashton, που κάνατε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Είμαι ευγνώμων που έχετε αναφέρει επανειλημμένα το θέμα. Η Αίγυπτος, η Αλγερία οφείλουν να κατανοήσουν ότι δεν θα συνεχίσουμε τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές αν δεν σεβαστούν τους ε, χριστιανούς. Το Σουδάν, ε, το Ιράκ ε, πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα δημιουργήσουμε ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών εάν δεν γίνει σεβαστή η ε, θρησκευτική ελευθερία στις χώρες αυτές. Πάρα πολλά βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν πρέπει να ενδώσουμε, γιατί αν ενδώσουμε, ε, δεν θα αναλάβει το δικό μας το έργο. Αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε επισκόπους από τη Μουσούλη, από τη Βαγδάτη. Οι επίσκοποι αυτοί απόψη με εμά. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε με αυτούς, σε αυτού αλληλεγγύη. Ε, πρέπει να είμαστε για μα το σημείο αναφορά, γιατί αλλιώ δεν θα είμαστε <clears throat> αξιόπιστοι. Αν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τους φίλους μας, τότε δεν είμαστε και αξιόπιστοι. Για ε, την ε, Ενωτική Αριστερά, Βερσά, για ένα, Βερζά, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η συνεδρίασή μας ε, φαίνεται να αναφέρεται τα μάλλα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υιοθετήσαμε σήμερα το πρωί την έκθεση Γκάλ και μία έκθεση για τα δικαιώματα των θυμάτων και μία για την εμπορία ανθρώπων ε, εδώ. Θα ήθελα να τονίσω την απόρριψη της ενίας ε, άδεια ε, για το γραφείο, για το βραβείο με συγχωρείτε Ζαχάροφ. Ήδη έχω τοποθετηθεί όμως και η έκθεση αυτή εντάσσεται στο ίδιο όραμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρουσιάζουν εδώ ορισμένοι συνάδελφοι και λυπούμε γι' αυτό. Είναι δύο ταχυτήτων. Εγώ σέβομαι την ε, ελευθερία ε, της ε, θρησκείας αλλά και την ελευθερία να πιστεύει κανείς ή να μην πιστεύει. Πάρα πολλοί άνθρωποι διώκονται στον κόσμο. Η συγκήτρια έχει αρνηθεί κάποιες τροπολογίες ε, σε σχέση με την ελευθερία της επίστης της θρησκείας ε, και της σκέψης. Γιατί δεκά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 ε, ε, παράγραφη για τους χριστιανούς και μόνο έξι παράγραφη για την ελευθερία της σκέψης γιατί αναφέρονται πάντοτε οι ίδιες χώρες η Ρωσία, το Ιράκ, το Ιράκ, η Λευκορωσία ή η Κούβα φυσικά ενώ δεν αναφέρουμε καθόλου σχεδόν την κατάσταση που έχουμε σε πολυάριθμες χώρες της Αφρικής και δεν αναφερόμαστε καθόλου στο Μαγκρέπ όπου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ε, πραγματικά διώκονται και στην Τινησία και στη Λιβύη και Λιβύη και τίποτα δεν και για την Κολομβία. Και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο. Πιστεύω ότι αν προσαρμόζουμε ε, τον ε, λόγο μας ε, ε, έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε και δρόμο να καλύψουμε και σας άκουσα κυρία Άστορ, με μεγάλη προσοχή. Για την ομάδα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας προβέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για το ότι δέχτηκε δικές μου πρωτοβουλίες για την θρησκευτική ελευθερία και τη συγχαίρω για την επιτυχία που σημείωσε κατά τη σύνταξη αυτή της έκθεσης. Όλο και πιο συχνά είναι τα τραγικά γεγονότα που αφορούν την ελευθερία των πιστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, έχουμε εμπόδια στην ελευθερία άσκηση θρησκευτικών ε, δικαιωμάτων. Αυτά γίνονται όλο και πιο συχνά. Και αυτές οι δολοφονικές πράξεις αφορούν τους πιστούς ε, όλων των ομολογιών, κυρίως τους χριστιανούς. Η θρησκευτική ελευθερία, κατά παράδοξο τρόπο, γίνεται ένα θέμα όλο και πιο λεπτό, αντί να είναι μία από τις πλέον φυσικές και αδιαμφισβήτητες ελευθερίες. Για όλους αυτούς τους λόγους, επαναλαμβάνω αυτό που έχω προτείνει και κατά το παρελθόν. Δηλαδή, να υπάρχει μία ειδική σχέση ε, που να είναι ετήσια ε, για να ελέγχουμε την κατάσταση των θρησκευτικών ελευθεριών ανά τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η έκθεση, η έκθεση ε, θα δίνει τη δυνατότητα ενδεχομένως και προληπτικών μέτρων. Ευχαριστούμε ε, για τους ε, μη εγγεγραμμένους. Σινκλέρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε γενιές παιδιών στα σχολεία της Σοβιετικής Ένωσης άκουγαν πως ε, ο Στάλιν ανακάλυψε τη μηχανή εσωτερικής ανάφλεξης. Εδώ οι Ευρωπαίοι έχουν μεγαλώσει ακούγοντας για την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι έχουμε κάνει όμως στην πραγματικότητα. Η συγγήτρια ε, υπογρυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πολλές προσπάθειες αλλά δεν δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι αποστολές στήρησης της ειρήνη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλέ, αλλά τι έγινε το 99 στο Βέλγιο με τον πρόεδρο Φερχόφστατ. Τι έγινε με την ε, εκδίωξη των ε, ε, Ρώμα από την, το από την Γαλλία φέτος. Την περασμένη εβδομάδα η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε ανησυχίες για την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προτεραιότητα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τι θα κάνουμε λοιπόν για όσους υποφέρουν παγκοσμίω. Την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή εγώ κατηγόρησα την Βελγική Προεδρία ότι είναι μια Προεδρία στενόμυαλη και κατά μεγάλη μου έκπληξη συμφώνησαν μαζί μου οι πρόσωποι τη Προεδρία. Φαίνεται ότι αυτό ακριβώ ήθελαν να είναι. Ήθελα λοιπόν η Βαρόνια Άστο να μου πει στην επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να παραστεί στι 10 Ιανουαρίου, ώστε να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων για το δίκτυο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία και να μα εξηγήσει ακριβώ τι σημαίνει για εκείνη η λέξη δράση. Ehm. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συγγεγραμμένους ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε με ε, Κατσμάρεκ για 1,5 λεπτά. Ο κύριος Κατσμάρεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Τρικένε για αυτή την έκθεση για τα ανθρωπίνα δικαιώματα το 2009 δεν ήταν ε, εύκολη υπόθεση γιατί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρήζει της προσοχής και της δεσμευσής μας. Στην ε, έκθεση πολλές φορές αναφερόμαστε στις ε, διάφορες χώρες και στους διάφορους οργανισμούς που πρέπει να αναλάμβουν δράση για να αυξήσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να επαληθεύουμε πιο συχνά αν ε, υλοποιούνται οι δεσμεύσει αυτέ. Και αυτό είναι το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαφορετικά, σε ένα έτο θα πρέπει να επαναλάβουμε πολλέ από τι σημερινέ παρατηρήσει. Έχουμε δίκιο όταν λέμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε οι κυβερνήσει των διαφορών χωρών ε, να σέβονται τι ε, ενδείξεις μας υποστηρίζω σε λέει η συγγήτρια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα πρέπει να υπάρχει μια γενική διεύθυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θα πρέπει να έχουμε και έναν υπατό εκπρόσωπο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο μήνυμα της έκθεσης. Αν μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό, τότε οι επόμενες εκθέσεις ε, ίσως ε, θα είναι ε, λιγότερο μακροσκελή και αυτή είναι η ευχή μα. Ευχαριστώ ο κύριο Τζάνικε για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνετε το λόγο. Σήμερα λοιπόν αναλύουμε μια ετήσια έκθεση η οποία ε, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι μια προσπάθεια το 2009 να αναλύσουμε κατά πόσον, το κατά πόσον ε, προστατεύτηκαν, ε, έγιναν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Κατά πόσον πέρυσι σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς η απάντηση δεν μπορεί να είναι καταφατική. Και επουδενή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόοδο στον τομέα αυτό το 2009. Αναφέρομαι στη θανατική ποινή, ε, στα βασανιστήρια σε πάρα πολλές χώρες. Ε, πονώ τη βία εις βάρος ε, των γυναικών, οι οποίες οδηγήθηκαν πολλές φορές σε εξαναγκαστική εργασία. Το ίδιο και τα παιδιά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αξίες μας είναι αδιαμφισβήτητες. Η μεγαλύτερη μας ανησυχία έγκυται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγωνιστεί περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ συμφωνώ με όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Αν όμως ε, ήταν... Ε, ε, μπορούσαν να εφαρμοστούν οι προτάσει μας, τότε πραγματικά θα είχαμε διαφύλαξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε Γκέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η έκθεση τη κυρία Αντρικέν ναι, είναι είναι το έγγραφο αναφορά. για όλα όσα λέγονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι καλό να μοιραζόμαστε διδάγματα με του εταίρου μα στον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ορισμένε χώρε είναι ακόμη στο μεσαίωνα σε ό,τι αφορά ε, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Ευρώπη θα εμπνεόταν ε, από ε, το να μην αγιοθετήσει μια ιδιαίτερα αλαζονική θέση κριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τι αρχέ των κρατών ε, μέλη των κρατών που συνεχίζουν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήταν ακόμη πιο αξιόπιστη αν τα 27 κράτη-μέλη δέχονταν ε, να εφαρμόσουν όλε τι αποφάσει του δικαστηρίου του Στρασβούργου που βρισκόμαστε εμείς δεν θα ήταν καιρός να έχουμε μια πιο επίσημη δέσμευση προκειμένου ε, να διασκεδάσουμε την παραμικρή αμφιβολία για την βούλησή μας να σεβαστούμε την αρχή των οργάνων που δημιουργήσαμε εμείς οι και Ευχαριστώ. Λοκμπίλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δυνατότητε ε, να βελτιώσει την κατάσταση σε πολλές χώρες. Είναι μια περιφερειακή δύναμη η οποία ε, θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να εφαρμόσουμε καλύτερη πολιτική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την υπηρεσία εξωτερική δράση έχουμε πλέον την ευκαιρία να σκεφτούμε το κατά πόσον η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποτελεσματικότητα που επιθυμούμε. Εγώ το εύχομαι αυτό και χαιρετίζω ε, το ότι αναθεωρείται η ε, πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που ανακοινώσατε εσεί, Βαρόνι. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι κατά πόσον όλα αυτά ε, θα μπορούν να βαδίζουν ε, παράλληλα και με την υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα ε, δημιουργήσετε εσείς στη δική σας την υπηρεσία. Γιατί υπάρχει ο φόβος ότι με τον τρόπο αυτό θα περιστούν περαιτέρω οι πόροι και δεν θα έχουμε πια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υπηρεσία υποσύσταση ε, τελικά θα είναι υπηρεσία φάντασμα αν δεν έχουμε ανώτατα κλιμάκια τα οποία να μπορούν να εκπροσωπήσουν την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, χρειαζόμαστε ένα ουσιαστικό, μια ουσιαστική ομάδα εμπειρογνωμόνων σε ανώτατο επίπεδο και ε, μετά μόνο τότε θα είναι δυνατόν να διοχετευτεί η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις ε, πολιτικές να γίνει mainstreaming. Θα ήταν ε, λοιπόν ε, αντιεπαγγελματικό και οπισθοχώρηση αν δίναμε ε, σημασία μόνο σε αυτή τη διάσταση του mainstreaming. Οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν περιμένουν μια άλλη διαφορετική πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μια απλή διοικητική αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τάνοκ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την κυρία Αντρικιάνια, την εισηγήτρια, για την ισόρροπη και πολύ λογική προσέγγιση που ακολουθεί στην έκθεση αυτή. Η ομάδα μου, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, οπωσδήποτε θέλει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι κάποιε φορέ τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αντισταθμιστούν και με τι ανάγκε τη Realpolitik. Διότι για ποιον άλλο λόγο θα είχε στατηγική εταιρική σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα, εκεί που θεωρούμε ότι οι ελευθερίε ε, που είναι θεμελιώδει δεν προστατεύονται αρκετά. Επίση, πρέπει να σκεφτούμε την ανθρωπιστική έχει προσφέρουμε σε αναπτυσσόμενε χώρε, αυτέ ακόμη που έχουν αξιολείπητη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω το Πακιστάν, οι γυναίκε και οι εκεί έχουν θεσμοθετημένη πλέον διακριτική μεταχείριση εναντίον του. Εδώ λοιπόν η έκθεση αυτή υπογραμμίζει την κατάσταση χωρών που για μένα θα ήταν ε, ιδιαίτερη ανησυχία, όπω η Κορέα, ε, το Βιετνάμ, η Ζιμπάμπου, η Βενεζουέλα, ε, και ε, άλλε. Στη Ρωσία επίση υπάρχουν ανησυχίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κεντρική ιδέα που διατρέχει την έκθεση αυτή είναι ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία έκθεση είναι στοιχεία που πρέπει να συμβαδίζουν. Όμω δεν έχω αμφιβολίε. Όταν αναφέρει το Διεθνέ Δίκαιο το Ευρωκοινοβούλιο για να καταγγείλει ε, την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν βασίζεται σε συγκεκριμένη ε, νομική βάση. Κένια και η Μαλαισία αναφέρονται αύριο σε ψήφισμα του Κοινοβουλίου ω χώρε που δεν σέβονται το Διεθνέ Δίκαιο. Πώ όμω νομικώ μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη στάση μα αυτή. Νομίζω ότι από αυτή, την, από αυτή την άποψη ε, πρέπει να αναλάβει δράση το θεσμικό σα όργανο. Σα ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριο Μπέλντερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Η δική μας δέσμευση για το σεβασμό των ε, κυρίων αποφασών του δικοστηρίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς και προσωπική εμπλοκή. Έτσι λοιπόν, ε, εδώ υπησέρχεται η έκθεση της κυρίας ε, Αντρικένε. Το σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι η ελευθερία θρησκευτική ε, πεποίθησης. Θρησκευτικές ελευθερίες αναφέρονται εδώ. Στις διπλωματικές σχέσεις θα πρέπει να ε, αναφερθούμε πάρα πολύ ε, συγκεκριμένα ε, σε αυτές τις σχέσεις. Έχουμε το χάρη έναν δικηγόρο στην Κίνα, ο οποίος εδώ και καιρό είναι υποκατοίκον περιορισμό και οι μυστικές υπηρεσίες τον παρακολουθών. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε και είπατε εκπρόσωπος να καταγγείλει το ζήτημα αυτό. Ας σκεφτείτε τον Τζαμπίμπη που ε, έχει καταδικαστεί σε θάνατο λόγω μιας ψεύδο βλασφημίας. Ε, το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ε, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, δηλώνει, πέρα από το να προβεί σε έρευνα βάσει το ισχύουσες νομοθεσία στο Πακιστάν για τη βλασφημία. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι θύνοντες θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά της κατάστασης αυτής. Κατόπιν έχουμε μία σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ισλαμικές Δημοκρατίες που πρέπει να καταγγελθούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Αντιπρόεδρε, έχουμε πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ, ο κύριος Μάλτσερ. Όταν ε, λέμε ή όταν η Κίνα λέει ότι πρέπει να ε, μποϊκοταριστεί ε, το Νομπέλ Ειρήνης και το Αφγανιστάν συμφωνεί, τότε για μένα αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πόσο δύσκολο είναι να ε, σεβαστούν οι μουσουλμανικές κυβερνήσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν ε, τις περιπτώσεις ε, διακριτικής μεταχείρισης ε, και μυσαλλοδοξίας έναντι των χριστιανών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και ανησυχίε στην Ευρώπη. Όλο και μεγαλύτερα προβλήματα σε μουσουλμανικούς κύκλους, εξαναγκασμό σε γάμο, η σαρία, αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά στην Ευρώπη. Εκείνο που πρέπει να καταδικάσουμε είναι αυτό ο πολιτιστικός σχέδιο. Ε, ε, που λέει ότι πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Ε, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ισότητα, στην ελευθερία και ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να περιοριστεί. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, λέει η Πρόεδρες, ότι ο κύριος Κούκαν ε, δεν είναι στην αίθουσα. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πρόντι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση Εντρίκενεν είναι μια θαυμάσια έκθεση συνολικά και επ' αυτής οι σοσιαλιστές και οι δημοκρατοί δούλεψαν πάρα πολύ για να τι αποδώσουν και ιδιαίτερη αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μία από τις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από την ώρα που συστάθηκε. Είναι ε, κάτι, μία απέτηση συνεκουανών και το Κοινοβούλιο πρέπει αυτό να το προβάλλει κάθε μέρο η παγκοσμιοποίηση και η αλλαγή της κοινωνίας μας επιβάλλουν ένα νέο όραμα διαφορετικό το οποίο απορρέει από, όλα αυτά που έχουν εθετηθεί μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εγγυηθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπάρχει ίση πρόσβαση στους ε, φυσικούς πόρους. Η κλιματική αλλαγή κατά τα επόμενα έτη θα προκαλέσει ένα τεράστιο αριθμό ε, προσφύγων από τις ε, πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Είναι λοιπόν καθήκον μας να συνειδητοποιήσουμε αυτές τις μεταναστευτικές ροές για να έχουμε τις κατάλληλες εκείνες πολιτικές που θα επιτρέψουν το σεβασμό ε, στην αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Ε, σήμερα δεν υπάρχει ο όρος ε, κλιματικός πρόσφυγας. Δικό μας καθήκον είναι να αντιμετωπίσουμε και την απερίμωση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα θέματα θελήσαμε να εντάξουμε στην έκθεση έτσι ώστε να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει Σακέ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και είπατε εκπρόσωπε. Αυτή τη στιγμή ε, είναι σημαντική μέρα για μας σήμερα. Γιορτάζουμε την απονομή του βραβείου Σακάροφ, όμως έχουμε και πολλά άλλα να κάνουμε πέρα από αυτό. Ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποια στοιχεία που αυτά είναι πολύ καλά συνταγμένη και ε, ισορροπή έκθεση. Η ανάγκη να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία μέσω τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και άλλων. Δεν είναι μόνο σημαντικό οι αυτούργοι να έρχονται ενώπιον τη δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα όσοι φοβούνται παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να παρατηρητέ, τουλάχιστον γίνονται ανεκτέ από κάποια αντιδημοκρατικά καθεστώτα, τότε να μπορούν του ε, υπεύθυνου για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να του κατηγορούν για τον πόνο που έχουν προκαλέσει και να του ε, ε, μπορούν να τους, να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους Ιρανούς λόγου χάρη που συστηματικώς ε, ασκούν λογοκρισία, ε, βασανιστήρια, παραβίαση των δικαιωμάτων των συμπολιτών τους, εκεί δεν έχει γίνει τίποτα. Και εδώ σίγουρα παραβιάζονται παγκοσμίω τα ανθρώπινα και τα οικουμενικά δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Βαντάλεν για 1,5 λεπτό. Κύριε Βαντάλεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε σε πολλά σημεία του κόσμου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βελτιωθεί. Σκεπτόμουν για παράδειγμα την Ανατολική Ευρώπη, κάποιες χώρες της Αμερικής. Ε, εδώ υπάρχει και μεγαλύτερη δημοκρατία, περισσότερη δημοκρατία μάλλον και περισσότερη σταθερότητα και ευημερία. Όμως υπάρχουν άλλες χώρες, όπως η Αίγυπτος, το Ιράκ, το Ιράν, το Πακιστάν, η Σομαλία και άλλε παρόμοιε, όπου οι χριστιανοί και μέλη άλλων θρησκευτικών ομάδων ε, δέχονται καταπίεση και διώξει. Βλέπουμε κατηγορίε ε, βλασφημιών να εξαπολύονται, ε, προσβολή θρησκευτικών πεπιθήσεων, υπάρχουν παρενοχλήσει, ε, ηλικιωμένοι και γυρεότεροι πέφτουν θύματα διακριτική μεταχείριση, μειονότητε και κοινότητε που έχουν ζήσει στι χώρε αυτέ για διάστημα μεγαλύτερο από οι ίδιοι μου αμεθανοί. Λοιπόν, Πρόεδρε, ένα, τουλάχιστον ένα στου πέντε ανθρώπου που διώκονται παγκοσμίω για τι θρησκευτικέ είναι χριστιανοί. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, κάτι περισσότερο, προκειμένου να ε, αντιμετωπίσουν αυτή τη θρησκευτική δίωξη. Ε, κυρία Άστον, τι σκοπεύετε να κάνετε από την άποψη των πολιτικών μέτρων για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σαλαβράκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε οφείλω να συγχαρώ την κυρία andrikien για την ολοκληρωμένη έκθεση που κατέθεσε. οφείλω να υπενθυμίσω σε όλους μας κύριε πρόεδρε ότι οι αρχαίοι έλληνες πριν από δύο χιλιάδες χρόνια είχαν πει πάντων μέτρων ο άνθρωπος. οι λατίνοι οι ρωμαίοι δύο αιώνες αργότερα είχαν πει homo hominis lupus ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος θέλω να δούμε κυρία πρόεδρε αν η ρίση των αρχαίων ελλήνων αποτελεί φιλοσοφική ρητορία ή εάν προχωρήσαμε. προχωρήσαμε σίγουρα πλην όμως δεν φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυστυχώς η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση που διακατέχει και έχει ξεσπάσει στην ευρώπη και στον κόσμο όλο έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και έχει πλήξει κατά κύριο λόγο τα φτωχά κοινωνικά στρώματα και τους έχει στερήσει ανθρώπινα δικαιώματα στοιχειώδους ε, αυτοσεβασμού. δεν θα πρέπει να μένουμε κυρία πρόεδρε και κυρία άστον ε, μόνο στα ρήματα μόνο στους λόγους. πρέπει να κάνουμε και πράξεις πρέπει να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα για την κοινωνική προστασία την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά κυρίως και την απασχόληση των νέων. υπενθυμίζω και πάλι η απασχόληση δεν είναι βιοπορισμός είναι δημιουργία αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας και συνθηκών ειρήνης μέσα στον χώρο της ευρώπης. σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Βέρτμαν, ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τον πολιτισμό δεν τον μετράει κανείς μόνο με την τεχνική πρόοδο και την ευημερία, αλλά όλο και περισσότερο με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτή η ρίση προέρχεται από μια εκπομπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τον 21ο αιώνα και πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για μας. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα δεν είναι κάτι το αυτονόητο και ε, όταν... Ε, μετράμε κι εμείς με διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Αυτό ε, ισχύει πράγματι και για την πολιτική μας κάθε πέμπτη απόγευμα θεσπίζουμε ψηφίματα, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν και πράξει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει σε όλου του τομεί τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζονται. Και εγώ είμαι υπέρ τη αναθεώρηση όλων των μέσων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα, γιατί προφανώ δεν είναι ότι λείπει η πολιτική βούληση. Εκείνο που λείπει είναι η εφαρμογή των αποφάσεων και των μέτρων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Μικολάζικ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Στον, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίες όπως η ισότητα, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μέχρι τώρα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχει και μία άσκηση συνεπού εξωτερική πολιτική με τη συνεισφορά των κρατών μελών. Η θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη πρόθεση τη δημοκρατία. Θα πρέπει αυτά να καταστούν τα κύρια στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής αλλά και όλων των ε, τομέων. Θα πρέπει τα ανθρωπίνα δικαιώματα να ενταχθούν ε, στην ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, το αν είχαμε και έναν ε, ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βοηθούσε να αυξήσουμε την ερωτότητα των ε, δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για το σημαντικό έργο της για την έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα έτη 2008 και 2009. Η έκθεση προσφέρει μια πλήρη εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο λόγο έχει ο κύριος Κάσμαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης ε, και την εισηγήτρια για την θαυμάσια έκθεση. Ε, Κυρία Άστον, χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα βρίσκεστε εδώ ε, διότι τελικά υποδεικνύεται ε, ότι δεν έχετε καμία, κανένα δισταγμό ε, να αντιμετωπίσετε εκείνου που του αφαιρούν ε, τη φωνή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα, είναι οικουμενικά. Η οικουμενικότητα όμως δεν ε, υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ε, συμφωνίες όπως με τις χώρες της Αφρικής και της Καρυβικής ε, όπου τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφιλοφίλων, των αμφιφιλοφίλων και των φιλομεταβατικών ποινικοποιούνται. Και γι' αυτό λοιπόν τι το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή διεύθυνση στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα. Ε, να ε, μπλέκονται βέβαια και με το εξωτερικό εμπόριο και τι εξωτερικέ υποθέσει, όπω είπατε και εσεί. Έχουμε συμφωνίε ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών, όπου το άρθρο 2 ποτέ κατ' ουσίαν δεν εφαρμόστηκε. Το Κοινοβούλιο υποβάλλει συστάσει ε, και φοβάμαι το Συμβούλιο τη αγνοεί. Έτσι λοιπόν θέλουμε να αναλάβετε την καθοδήγηση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε σχέση. Το 2009, σας συγχαίρω, ε, το Συμβούλιο ενέκρινε ε, το TOCET, ε, την πλατφόρμα αυτή των λεσβιών και των φιλομεταβατικών, των αμφιφιλοφίλων. Εγώ λοιπόν σας εμπιστεύομαι. Αυτό ήθελα απλά να εκφράσω. Ευχαριστώ. Μακμίλαν Σκότ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ μιλώ ως, προς, ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρωπινά Δικαιώματα και ευχαριστώ την συγκεκριμένη την εξαιρετική έκθεση η κυρία Στον στην ομιλία τη. Μίλησε για τις νέες δομές στο ιστορικό της υπηρεσίας ε, όταν εγώ έμαθα ότι το, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα, θεώρησα ότι είχαμε μια δομή για το σοβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία. Εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά κυρία Άστον είπε ότι η Κομισιόν ήθελε να ε, το καταργήσει τώρα η κυρία Άστον δεν μίλησε για mainstreaming στο λόγο της όταν μιλά ε, για τις ε, ε ε, ουσιαστικά εδώ βλέπουμε μια εξωτερική πολιτική που όμως θα πρέπει ε, να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα χρειαζόμαστε ίσως και έναν ειδικό εκπρόσωπο όπως και ο κύριε Χάτολα και εγώ ε, θέλω να τονίσω το εξής. Χίλια άτομα περίπου είναι ενωμένα σε όλο το, πέρα από τον Ατλαντικό στο Όσλο έχουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, ε, και άλλους φορείς ε, και όλοι όμως είχαν μια ενωμένη προσέγγιση ως ενωμένη κοινωνία των πολιτών στο μέλλον. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί αυτή την soft power θα πρέπει να προωθεί και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε το λόγο Πορέμπα για ένα λεπτό. Ο κύριος Πορέμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε. Πράγματι η έκθεση της συναδέλφου Αντρικέν είναι ιδιαίτερα διεξοδική. Ε, νομίζω ότι καλύπτει όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2008-2009. Μιλά για την διακριτική μεταχείριση κατά των ε, χριστιανικών ομάδων, όχι μόνο σε τρίτε χώρε αλλά και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πολιτικά εργαλεία και διπλωματικά μέσα για να αναχαιτήσει αυτό το είδο τα φαινόμενα. Ε, ε, μπορεί να καταδικάσει με τρόπο κατηγορηματικό και αποφασιστικό τέτοιου είδου ε, διακρίσει. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση και σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Η Συμφωνία Συνεργασία με τη Ρωσία, ε, που ε, ήταν πρόσφατα αντικείμενο διαπραγματεύσεων, είναι μια περίφημη ευκαιρία για να μπορέσουμε να τονίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό διεξοδικά. Να μην ξεχνάμε όσο είναι θύματα διακριτική μεταχείριση στη Ρωσία, πολιτικών διώξεων και ακόμη και επιχειρηματίε ε, οι οποίοι διώκονται ε, και αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί πολλές φορές απλώς έχουν την τόλμη να ζητούν την αλήθεια για το πώς λειτουργεί το κράτος τους. Ευχαριστούμε. Το λόγο ο κύριος Κάμπελ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ενώ όλοι ενώνουμε τι φωνέ μα για να καταδικάσουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρε όπω το Ιράν και η Κίνα, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάποια διάκριση για το τι συμβαίνει ε, με την βιομηχανία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, κατά πόσον υπάρχει μία έξαρση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουμε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ε, κάποιες φορές ε, υπερβαίνει τα εσκαμμένα, υπάρχει υπερβολική υπερβολικές, ε, υπερβολικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, ε, υπάρχουν ε, νόμοι παράνομοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου για κάποιους παρανόμους διαμένοντες τα δικαιώματά τους προστατεύονται καλύτερα από ότι των νομίμων κατοίκων. Έτσι λοιπόν η ρήτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάποιες φορές φαίνεται να δημιουργεί ένα βαθύ πρόβλημα με τη συμμετοχή δικηγόρων, τρομοκρατών και δημοσιογράφων οι οποίοι όλοι μπορούν να εκφράσουν ανεπιστήμα εμπόδιστα την απληστία του. Αυτό πρέπει να ε, πάψει. Ευχαριστούμε το λόγο ο κύριος Ομπερμάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει περισσότερο. Η έκθεση αυτή αναφέρει σωστά την ε, διακριτική μεταχείριση κατά των χριστιανών. Αυτό το βήμα το βρίσκω θετικό. Απλώς να δώσω κάποια παραδείγματα Κάποιε φορέ υπάρχουν βίε ενέργειε κατά των χριστιανών στην Αίγυπτο, την Τουρκία στην, ε, και σε άλλε χώρε και δίνουν μάχη για την απλή σωματική του επιβίωση. Πρέπει να από τι χώρε αυτέ λοιπόν να είναι πιο ανεκτικέ. Αυτό λοιπόν ε, θα προκαλούσε μεγάλο κόστος χωρίς αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν αρκετά μέτρα πίεσης. Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Καμία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπάρχει ροή κονδυλίων χωρίς την διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των μειονοτήτων, κυρίως ε, των χριστιανικών μειονοτήτων. Κυρίες και κύριοι, τα επιχειρήματα πρέπει να είναι πιστικά ε, και νομίζω ότι το να ασκείται πίεση είναι πιο αποτελεσματικό όταν δεν βοηθούν τα ανθρωπιστικά ε, επιχειρήματα. Γκάλ για 1,5 λεπτό. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τη συναδελφό μου την κυρία Αντρικίνη για την εξαιρετική δουλειά της. Ε, είδαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τροπολογιών που κατατέθηκαν και αυτό μας έδειξε πόσο Ηράκλειος ήταν ο άθλος της. Χαίρομαι πάρα πολύ που στην έκθεση δίνεται έμφαση στις ε, πιο ευάλωτες ομάδες και που χρειάζονται περισσότερο προστασία όπως ε, οι ηθαγενείς, οι εθελοντικές μειονότητες και τα παιδιά. Πιστεύω ότι τα μηνύματα μας ε, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο για την εξωτερική υπηρεσία, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τα καθήκοντά της ε, έγιναν αποδεκτά με ανοιχτό πνεύμα. Νομίζω ότι οι προσπάθειες της κυρίας Άστον θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις πολιτικές. Αυτό θα είναι μία από τι κύριε δραστηριότητε τη Υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δρούμε πιο συντονισμένα στις εξωτερικές μας σχέσεις και θα πρέπει να σεβαστούμε το πνεύμα όσων υιοθετήσαμε για να μην διακινδυνεύσουμε την αξιοπιστία μα. Πρόκειται για μία συζήτηση η οποία γίνεται άπαξ της στην Ολομέλεια και αν δούμε το έγγραφο, ε, βλέπετε ότι προσπαθούμε εδώ να περάσουμε ένα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφύγουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Υπέτη Πρόσωπε, είμαι πολύ ικανοποιημένος που τα ανθρώπινα δικαιώματα εντάσσονται στα ε, καθήκοντα τη υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την υπεράσπιση του σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι μέλος τη αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Ρωσία και χαίρομαι επειδή στην έκθεση αυτή έχουμε παραγράφους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Αναφέρονται διάφοροι υπερασπιστές ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η υποστήριξη από τις ε, Βρυξέλλες και από το Στρασβούργο για τα άτομα αυτά είναι θεμελιώδης έτσι λοιπόν ε, πιστεύω ότι χρήζουν της δικής μας υποστήριξης πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στα άτομα αυτά και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και απευθύνω έκκληση στην κυρία Άστον. Ευχαριστώ, Σόνικ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση για την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το 2009, η έκθεση αυτή συμβαδίζει με μια ε, λυπηρή πραγματικότητα. Ο Λουί Ξιάομπο που είχε κερδίσει το βραβείο Νομπέλ και άλλοι άνθρωποι και ο κύριος Φαρίνιας δεν ε, έλαβαν ε, το δικαίωμα, το δυνατότητα να ταξιδέψουν. Συναντηθήκαμε με επισκόπους από το Ιράκ και μας είπαν ότι εξακολουθούν να είναι μάρτυρες διωγμών των χριστιανών. Υπήρξαν επιθέσεις στον καθεδρικό ναό στη Βαγδάτη. Άρα δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε πρόβλημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου ανάλογη θα πρέπει να είναι και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωση. Εγώ ε, προσυπογράφω αυτά που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Μπούζεκ, που ανέφερε ότι η επίθεση κατά των χριστιανών στο Ιράκ θα πρέπει να είναι για μας προτεραιότητα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι πολίτες αυτοί να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η μόνη ιερατική ε, σχολή που υπάρχει σε αυτή τη χώρα έκλεισε. Η συνθήκη της Λισαβόνας από τότε που ετέθη σε ισχύ υπάρχει πλέον ελπίδα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει όμως να δραστηριοποιηθούμε σε διεθνή διεθνές επίπεδο και γενικότερα ε, να βελτιώσουμε την ασφάλεια που υπάρχει ε, ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει επόμενη ομιλητρία, ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ω Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ανάπτυξη, εγώ ασχολούμαι με τα προβλήματα πολλών κρατών, κυρίω ε, στην Αφρική, όπου ε, καταπατώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλέ φορέ μάλιστα ξεχνιόνται και τελείω. Την ε, προηγούμενη Κυριακή γύρισα από μια επίσημη επίσκεψη στο Κονγκό, όπου εκτό από τι θεσμικέ επισκέψει ήθελα να έρθω σε επαφή και με εκπροσώπου των ΜΚΟ που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και με νύχια εξ αυτών δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Συνάντησα ε, τα θύματα σε μια χώρα όπου ο βιασμός θεωρείται όπλο ε, του πολέμου. Έχουμε λοιπόν μαζικούς βιασμούς και άλλες, ε, άλλα συστηματικά εγκλήματα κατά της κοινωνίας, εγκλήματα κατά των γυναικών και των μωρών, των παιδιών κυρίως. Έχω λοιπόν αυτή την πρόσφατη εμπειρία. Όμως η έκκληση που θέλω να απευθύνω αφορά την αναγκαιότητα να καταδικάσουμε ε, κατηγορηματικά τα εγκλήματα εις βάρος των γυναικών. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να δίδει περισσότερα κονδύλια στις πρωτοβουλίες για την προστασία των γυναικών από το βιασμό και από άλλες μορφές άσκησης μορφής βίας, όπως παραδείγματος χάρη τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων. Γιατί και αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως όσον αφορά την φύση της γυναίκας. Ευχαριστούμε, κύριε Ματέρα, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, λέει Άστον, συνάδελφοι, η δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, εκπροσωπεί μια ιστορική ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε σοβαρά ζητήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ιδιαιτέρω θα πρέπει να αναλάβει, να, να προωθηθεί ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό να βρίσκεται στο κέντρο των διαφόρων ε, τυχόν τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των πρεσβειών των κρατών μελών, με τον κοινό σκοπό να υιοθετηθεί μια στρατηγική αναχώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι οι ιδιαιτερότητε τη κάθε χώρα είναι πολύ αξιοσημείωτε μεταξύ των διαφορών χωρών. Η θανατική ποινή, λόγου χάρη, που σε διάφορε περιοχέ του κόσμου ισχύει, είναι από τι πιο απάνθρωπε μορφέ ε, εφαρμογή του νόμου. Και προκαλεί σοβαρέ ανησυχίε το γεγονό ότι παραμένει αυτή η θανατική ποινή στη Λευκορωσία, τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα που την εφαρμόζει ακόμη. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να πάυσει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, των οποίων, τις οποίες είναι οι θύματα γυναίκες, όπως η κλητεροδεκτομή. Και όλες οι δικές μας πολιτικές θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ε, ε, ακολουθούν τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου ζητείται διεθνής, μορατόριο για τον ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων των γυναικών. Εδώ λοιπόν και κλείνω πρέπει να, εντατ να εντείνουμε τις προσπάθειες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ώστε να ε, είναι πιο εντελεχής η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Ξεκινούμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 15 αγορητές. Δεν ξέρω εάν θα μπορέσω να δώσω χρόνο σε όλους. Όμως ξεκινούμε με τον κύριο Σόμπορ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι παρά το ότι σε πολλούς τομείς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είδαν παραδειγματικά σε δραστηριότητες ένταξης. Υπάρχουν κάποιες χώρες ε, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται ε, σε σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε καθυστερήσει. Θα ήθελα να καλέσω τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και το ΟΗΕ καθώς και τα προοδευτικά πρωτόκολλα. Επίσης, ε, θέλω να μιλήσω για την προστασία των εθνοτικών ε, μειονοτήτων και τη σχετικής σύμβασης, όπως και της ε, Ευρωπαϊκής Χάρτας για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για το μέλλον του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτές τις συμβάσεις. Πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τις δραστηριότητές μας στους διεθνείς οργανισμούς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εγγυθούμε την πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κόπα, κυρία Κόπα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπεια στι αρχέ και αξίε τη, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Έχουν όμω πολλά να γίνουν και η συνθήκη τη Λισαβόνα έρχεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μα στον τομέα αυτό είναι πεποίθηση όλων μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ότι πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. η σωστή εφαρμογή των εργαλείων που ήδη υπάρχουν μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο για την προστασία τους. σε υψηλή προτεραιότητα πρέπει να τεθεί η επικύρωση όλων των διεθνών συνθηκών ενάντια στα βασανιστήρια και κάθε άλλης μορφής απάνθρωπης μεταχείρισης η συμπερίληψη της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες αλλά και η παρακολούθηση της εφαρμογής είναι ουσιαστικά μέτρα και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά. ειδική αναφορά νομίζω πρέπει να γίνει στην ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέρο τη συζήτηση μα σήμερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι εξωτερικέ και εσωτερικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι και η κατάσταση των γυναικών. Και ήθελα εδώ να σταθώ, ιδίω στι περιοχέ όπου υπάρχουν σειράξει, στο Κονγκό, στη Γάζα και στο Ιράν. Τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει πλέον να τα παραμερίζουμε και να τα παραβλέπουμε. Οι γυναίκε ε, πολλέ φορέ αναγκάζονται να υποστούν τι χειρότερε συνέπειε από τι καταστάσει των εχθροπραξιών και τη σύγκρουση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν αυτή την πλευρά, αυτή την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατάσταση των γυναικών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζεται τα συμφέροντα των γυναικών στην εξωτερική τη πολιτική και την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάσταση των γυναικών, οι συνθήκε διαβίωση του σε ένα μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών πολλέ φορέ ε, θυσιάζονται ε, στο όνομα των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να ζητούσουμε να προβλεφθούν συγκεκριμένα και χειροπιαστά βήματα, ώστε οι αρχέ γενικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφραστούν σε συγκεκριμένε δράσει. Συγκεκριμένε δράσει που να προτείνουν ε, την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ευχαριστούμε. Λούνατσεκ. Δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, όταν ε, βλέπουμε κυβερνήσεις όπως η Γαλλική και η Πορτογαλική να αποκλίνουν ε, από εδώ είμαι. Όταν κυβερνήσει όπω η Γαλλική Περνιστή ε, αποκλίνουν, μάλλον υπάρχουν τεράστιε διαδηλώσει ε, ε, και προσπαθούν να τι κρύψουν για όταν ε, επισκέπτονται κάποιοι Κινέζοι ηγέτες και προσπαθούν να το κρύψουν. Τι να σας πω, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε με μία και μόνη φωνή. Τώρα, επειδή εσείς από την πλευρά του Συμβουλίου, ποια είναι ε, η φιλοσοφία πίσω από αυτή την επιλογή. Επίσης, ε, οι ίδιοι μας ευρωπαϊκοί διπλωμάτες θα ήθελαν να έχουν ως προτεραιότητα ε, τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό δεν αποτελεί παρά τρίτη ή τέταρτη προτεραιότητα και όχι πρώτη. Η διπλωμάτες μας ε, θα πρέπει καθημερινά να έχουν στο επίκεντρο το έργο του το έργο τους ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια διεύθυνση ειδική που να ασχολείται με το θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, το λόγο συνάδελφος Μπρόνς. Όταν ακούσαμε από τον κύριο Φορίνιας για την Κούβα σήμερα το πρωί εντυπωσιάστηκα ότι μίλησε για τον εαυτό του και για τους συναδέλφους του ότι είναι μια μη βίαιη αντιπολίτευση στην Κούβα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τα δικαιώματα ανθρώπων που ε, δεν είναι βίαιοι ε, και ούτε και δέχονται τη βία. Οφείλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι σε ορισμένε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες διώκονται γιατί ε, είναι αντιφρονούντες όπως ο κύριος Βίλντερς στην Ολλανδία. Οι απόψεις για ακαδημαϊκά ε, θέματα, χωρίς όμως άσκηση βίας. Ε, πολιτικά κόμματα χωρίς βίες ε, διασυνδέσεις απαγορεύτηκαν στο Βέλγιο και μια τέτοια παρεμφερής προσπάθεια απέτυχε στη Γερμανία γιατί αποδείχθηκε ότι τα στοιχεία είχαν μαγειρευτεί από μυστικούς πράκτορες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης και εκεί υπήρχε μια τέτοια προσπάθεια με στόχο να κλείσουν την έκφραση μιας πολιτικής άποψης. Για κολλήνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέντι ε, Άστον, η πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, είναι πλέον σε μια καμπή. Η κυρία Αντρικένεν πρέπει να στηριχτεί και κατέστησε απόλυτα σαφές ε, πόσο σαφείς πρέπει να είμαστε. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί αποτελεσματικά να αναπτύξει τις δράσεις του δείχνοντας και κάποια ευαισθησία απέναντι στα κράτη-μέλη και υπολογίζοντα την ευαισθησία αυτή. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια σαφής πολιτική. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα άμεσα, τα δικαιώματα των νέων, των γυ γυναικών, των αναπήρων που έχουν μια ειδική θρησκευτική προσέγγιση ε, και ε, διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Ο καθένας να μπορεί ελεύθερα να εκφράζει τις απόψεις του. Σήμερα λοιπόν ε, πάρα πολύ σημαντικές διατάξεις θεσπίστηκαν από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε μόνο μέσα από τον ισχυρό διάλογο με τρίτες χώρες θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά αμυγός και μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρονικόλας. Κυρία Άστον, είναι με ιδιαίτερη χαρά που ακούει κανείς την κατεξοχήν υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνει απερίφραστα ότι είμαστε υπέρ της εφαρμογής των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ως ευρωπαϊκή ένωση έχουμε να συνεισφέρουμε τα μέγιστα για την εφαρμογή αυτών των αρχών και ελευθεριών που είναι κοινά για όλη την ε, οικουμένη ούτως ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αυτό το θετικό ρόλο. γνωρίζετε τις θέσεις μας ότι αποζητούμε να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο τμήμα για τα για τι ανθρώπινες ελευθερίες πολύ περισσότερο να υπάρχει μια εποπτεία και να υπάρχουν απεσταλμένοι. θα έλεγα όμως κυρία Άστον, ότι οφείλουμε εκτός από τα εκτός να δούμε και τα εντός και προερχόμενος από την κύπρο θα έλεγα ότι έχουμε χιλιάδε πρόσφυγες ελληνοκύπριου που στερούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους πρόσβαση στο σπίτι τους όπως επίσης έχουμε μια τουρκοκυπριακή κοινότητα η οποία καταδυναστεύεται από την τουρκική κατοχή. οργανώστε το τμήμα σας μια συμβουλή και μια παράκληση στείλτε τον πρώτο σας απεσταλμένο στο έδαφος της κυπριακής δημοκρατίας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σμιτ. Χωρίς μικρόφωνο. Ζητώ συγγνώμη. Θα ξαναρχίσω. Νομίζω ότι ο David, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο David Ισακ ακόμα βρίσκεται στη φυλακή και δεν έχει δικαστεί. 2.317 μέρες είναι κρατούμενος και όσον αφορά τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έπρεπε να μπορέσουμε να δράσουμε αμεσότερα, ακόμα και εάν υπάρχουν παραβάσεις εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέβη Άστον, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση στην Ερυθρέα, έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο Ντέιβιτ Ίσακ. Θα πρέπει να το λάβουμε πιο σοβαρά πλέον το θέμα και να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση της Ερυθρέας. Όλες οι διαπραγματεύσεις με την Ερυθρέα θα πρέπει να υπόκεινται στην ελευθέρωσή του. Βασίζομαι σε εσά και πιστεύω ότι θα το καταφέρετε, λέει, Άστον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρζίπ. Ο κύριος Τζίμπ, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Αντρικένε για την έκθεσή της και παράλληλα θα ήθελα να δηλώσω ότι αφότου ετέθησε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας ισχύει μια νέα κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα διότι θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίζεται και η εμπορική μας πολιτική. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τη σημερινή απονομή του βραβείου Ζαχάροφ βλέπουμε ότι πολλές φορές εισακούνται τα αιτήματά μας. Πολλές φορές διώκονται χριστιανικές μειονότητες ανά τον κόσμο και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με το, ε, με τα Ηνωμένα Έθνη, με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και σε πολλά κράτη-μέλη, διότι υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα για το πώς ε, και τι επιπτώσεις υπάρχουν ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Thank you, Madam Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Λέβη Άστον. Παρότι η έκθεση ε, εμπεριέχει πολλά σημαντικά θέματα, θα ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το θέμα του Σεργέη Μακνίσκη. Η στρατηγική του είναι παρόμοια με άλλε αντίστοιχε περιπτώσει που δεν τι έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμή. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στι ρωσικέ αρχέ ότι τέτοια γεγονότα θα πρέπει να διερευνηθούν όπω προβλέπει και η αρχή του κράτου δικαίου. Αντί ανταυτού, οι, οι ερευνητές ε, και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το θάνατο του ανθρώπου αυτού αγνώρισαν πολλά γεγονότα. Ε, πρόκειται για κακο, κακή εφαρμογή της δικαιοσύνης και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια ε, σε τέτοιες ε, περιστάσεις. Θα πρέπει να μην ξεχνάσουμε τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σας ενθαρρύνω, συνάδελφοι, να υποστηρίξετε την αντροπολογία 25 που προτείνει να υπάρξουν κυρώσεις για 60 Ρώσους αξιωματούχους που έχουν εμπλακεί στην ε, υπόθεση αυτή μέχρι να χυθεί το φως ε, στις ε, συνθήκες θανάτου του ανθρώπου αυτού στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο κ. Προτάσφιτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλο τη Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ω μέλο τη Επιτροπή αυτή θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Ανδρικίενε ε, για την καλή ε, έκθεση. Ω πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία ε, για τη σχέση με τη Λευκορωσία, χαίρομαι για την κατάσταση στη χώρα αυτή, αν λάβουμε υπόψη το πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα Υπάρχει πρόβλημα με τις εθνικές μειονότητες και πρόβλημα ε, του συνέρχεστε. Επίσης χαίρομαι για την αναφορά ε, περί περιστολής της πρόσβασης ε, στο ίντερνετ. Η Λευκορωσία δυστυχώς είναι ένα τέτοιο θλιβερό παράδειγμα. Θα ήθελα η Λέδη Άστον να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της Λευκορωσίας να ασκήσει πίεση σε αυτούς που θέλουν ε, να μειώσουν την ελευθεροτυπία. Η κυρία Άουταλα, Χάουταλα, συγγνώμη. Ε, Θα ήθελα, Πρόεδρε, να θίξω ένα ζήτημα το οποίο θίγει και από άλλους συναδέλφους. Δηλαδή καταστολή των δικαιωμάτων των ε, χριστιανών. Θα ήθελα για να υπάρχει μια συνέπεια οι συνάδελφοι να ενδιαφερθούν και στην ε, καταστολή δικαιωμάτων άλλων θρησκειών διότι μας λένε άλλες χώρες ότι είμαστε μονομερείς και μεροληπτικοί και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι. Θα ήθελα λοιπόν κατευθυντήριες ε, γραμμές της κοινή ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορά όλες τις μειονότητες και τις ε, θρησκείες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Βαρόνι Άστον, θα απαντήσετε για τις νέες ανθρωπιστικές, τη νέα ανθρωπιστική διάρθρωση που θα υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών ε, Υποθέσεων Εξωτερικής Δράσης που θα αρχίσει να λειτουργεί τις επόμενες εβδομάδες. Δίνουμε το λόγο στην ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Άστον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για όλες ε, τις παρεμβάσεις στον, ε, στη συζήτηση αυτή που βρήκα πολύ ε, χρήσιμες. Σήμερα είμαι στην πλευρά του Συμβουλίου, νωρίτερα ήμουνα στην πλευρά της Κομισιόν. Φροντίζω να κινούμε ανάμεσα στους δύο αυτούς φορείς. Να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Αντρική θερμά για την δουλειά που έχει κάνει και να την συγχαρώ για την έκθεσή της, η οποία είναι πολύ χρήσιμη. Θα μου επιτρέψετε την απάντησή μου να τη χωρίσω σε τρεις ομάδες. Θα ξεκινήσω από το θέμα που έθιξε η κυρία Χάουταλα στο τέλος και που ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι. Καταρχήν να είμαι απόλυτα σαφής. Εγώ μιλάω για mainstreaming διότι πολύ συχνά στη ζωή μου είδα τις τα ανθρώπινα δικαιώματα να εγκαταλείπονται στην ε, άκρη ενός ε, οργανισμού ε, και να εξετάζονται παρεμπιπτόντως με τρόπο που δεν πρόκειται να οδηγήσει σε καμία διαφορά. Ε, δεν λέω ότι το κάνει, αυτό, το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά θέλω να φροντίσω να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όταν ολοκληρωθεί η δομή, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ε, θα φροντίσουμε να αναγνωρίζονται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα φροντίσουμε να έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη που ζήτησαν οι συνάδελφοι εδώ. Δεν θέλω όμω τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι ένα θέμα εγκαταλελειμμένο σε μια γωνία. Θέλω να είναι ε, ε, ε, ένα ασημένιο νήμα συνδετικό, ισχυρό που να λάμπει και να φαίνεται από όλου. Αυτό θέλω να πετύχω κατά τη διάρκεια τη θητεία μου και ε, είμαι αφοσιωμένη ε, ε, κατά 100% στον στόχο αυτόν. Είναι κάτι που θα απαιτήσει χρόνο και θα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε τόσο καλά όσο θέλω, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει να το κάνω και με ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο να καταλάβει τι θέλω να κάνω. Και θέλω να φροντίσω η ευθύνη καθενός να είναι το θέμα αυτό. Ναι, θα πρέπει να παρακολουθείτε, ναι, θα πρέπει ε, να υπάρχουν υπεύθυνοι, αλλά δεν θα είναι ε, ευθύνη κάποιων λίγων, είναι ευθύνη όλων μας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα δείτε πολύ σύντομα της, ε, την δομή, συμπεριλαμβάνεται, θα το δείτε σύντομα. Όσον αφορά τους προέδρους ε, των ομάδων εργασίας, ε, θα ε, κανονίσουμε σύντομα συναντήσεις. Θα ορίσω τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα δούμε αν αυτός θα έχει θέση στο, στις Βρυξέλλες ή στις, ή σε άλλες πρωτεύουσες. Κατά ε, τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ε, υπήρχε μια μονάδα που είχε να κάνει, ε, υπήρχε μια ενότητα που είχε να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ δεχτείτε ότι αποτελεί τον θεμελιώδη πυρήνα της δομής και είμαι αποφασισμένη να αποτελεί, να αποτελεί το πράγμα αυτό ευθύνη όλων. Ε, επόμενο θέμα είναι η ευρύτητα των θεμάτων. Δέχομαι αυτά που είπαν διάφοροι για την θρησκευτική πίστη. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, αυτό συζητήθηκε και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αυτή την εβδομάδα. Και έχουν δίκιο οι συνάδελφοι, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα γυναικών, παιδιών, ε, ε ομοφιλοφίλων ε, και άλλων. Ε, το για να εφαρμόζονται σε κάποιον τα ανθρώπινα δικαιώματα αρκεί το να είναι άνθρωπος. Αυτή είναι η προσέγγιση μας εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους. Το τρίτο που θέλω να πω έχει να κάνει με αυτά που βλέπουμε ότι ξεκινούν να γίνονται και όπου συμμετέχουμε εμείς. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, φέτος ε, ε, οδήγησε σε τέσσερα κράτη να αναγνωρίσουν το καταστατικό του. Εδώ παίξαμε κάποιο ρόλο. Εγώ έχω στείλει προσωπική επιστολή στον Πρωθυπουργό κάθε κράτος που δεν έχει επικαιρώσει το, το, το δικαστήριο και ως ανταπόκριση στην επιστολή αυτή είχαμε τα τέσσερα αυτά τα γράμματα. Ε, ε, ε, είχαμε την επικύρωση των τεσσάρων των χωρών. Επίσης, πυρηνικό μέρος της δουλειάς μας είναι αυτό και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Πρώτον, λοιπόν, σημαντικό είναι ο κόσμος να μάθει τι είναι αυτό που κάνουμε. Δεύτερον, να καλύπτουμε όλους και Τρίτον, να φροντίσουμε ε, να δούμε πού μπορούμε να οδηγήσουμε σε αλλαγή της κατάστασης. Και ε, στην, μεταρρύθμιση, στην αναθεώρηση θα πρέπει να εξετάσουμε τρόπους ε, πρακτικούς και καιροτόμους να περάσουμε το μήνυμά μας. Θέλω να είμαι δημιουργική στην εργασία μας που κάνουμε ε, επιτόπου με τους ανθρώπους. Ε, θέλω να είμαστε καινοτόμοι και δημιουργικοί ε, κατά την εξέταση τρόπων να θέσουμε εκ νέου το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 27 κράτη-μέλη έχουμε. Είναι λοιπόν σημαντικές οι δηλώσεις που κάνουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ανταποκριθούμε όσο γίνεται περισσότερο στις ανησυχίες ε, ατόμων, ε, οργανισμών και να οδηγήσουμε σε πραγματική αλλαγή της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Άστον. Η κυρία Αντρικέ είναι η συγγήτρια, είναι η τελευταία που παίρνει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου είπαν ότι δεν ήταν ακριβής η αγγλική διερμηνία της ε, ομιλίας μου. Λυπάμαι γι' αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, μετά από αυτή τη συζήτηση θα μεταφράσω εγώ η ίδια την ομιλία μου στα αγγλικά και θα την στείλω σε όλους τους συναδέλφους, ε, καθώς και στην ύπατη εκπρόσωπο. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ε, σημερινή συζήτηση για τη θετική τους αξιολόγηση και για τις ε, παρατηρήσεις τους, που είναι επίκαιρες για το συνάδελφο που μίλησε για τι ε, χριστιανικέ μειονότητες σε διάφορες χώρες, ε, λέγοντας ότι το θέμα αυτό δεν το αντιμετωπίζει, δεν το εξετάζει η έκθεση, θα ήθελα να σας ε, παραπέμψω στην παράγραφο 126. Υπήρχε και ένα κεφάλαιο που μιλούσε για την θρησκευτική ελευθερία και για τις χριστιανικέ χριστιανικές θρησκευτικές οι οποίε αναφέρονται και σε συγκεκριμένες παραγράφους. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, Βαρόνια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ελέγχει το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και θα συνεχίσουμε να επικρίνουμε την αδράνεια ή την αναποτελεσματικότητα των δράσεων που, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη φετινή έκθεση τονίζουμε ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκάθαρους στόχους και ορόσημα για να δούμε ε, πώς, πώς αποτελέσματα φέρνουν οι δράσεις μας στον τομέα της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε εκφράσει την απογοήτευσή μας για την έλλειψη πρόοδου σε ό,τι αφορά τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαβουλεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λεδιάστον ε, έχει συμφωνήσει μετά από μεγάλες προσπάθειες για τα πιο κρίσιμα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δείχνει ότι είναι ενωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση της δημοκρατίας, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Επίσης δείχνει ότι οι μέρες όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς χειροκροτούσε την Κομισιόν ε, και το Συμβούλιο έχουν παρέλθει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα είναι σημαντικός και σοβαρός εταίρος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα πραγματικότητα αυτή. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Αντρικίνε. Ε, τελείωσε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο ε, το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Μια μικρή ανακοίνωση πριν περάσουμε στην επόμενη συζήτηση. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι η κυρία Πασκά